Λοιπόν, σα παρακαλώ, περιμένω να επανελθούν στι θέσεις. Μία ανακοίνωση όσον αφορά την απόφαση διαφόρων επιτροπών να ξεκινήσουν οι διαθεσμικέ διαπραγματεύσεις με εφαρμογή του άρθρου 69.4, παράγραφο 1, που αναγγέλθηκε, αναγγέλθηκε στην ε, συνεδρίαση τη Δευτέρα. Ζήτησα αιτήματα ψηφοφορία με βάση το άρθρο 69 σε παράγραφο 2 από τι ομάδε Γκουέντζιελ, Άλντε, EFTD και ECR για την απόφαση της Επιτροπής Κιούλτ να ξεκινήσουν οι οργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τις έκθεσεις για τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Για την ε, αλλαγή της πραγματικότητας αγοράς είναι η έκθεση Φερχάιεν Κάμερβερτ. Η ψήφιση, η ψηφοφορία για την απόφαση της Κιούλτ να ξεκινήσουν οι οργανικές διαπραγματεύσεις θα γίνει αύριο. Όσον αφορά τις αποφάσεις των Επιτροπών ΙΝΤΑ, ΙΤΡΕ, ΙΜΚΟ, ΠΕΣ και ΛΥΜΠΕ για να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσει, δεν έλαβα κανένα αίτημα ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Αυτέ οι επιτροπέ μπορούν λοιπόν να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει. Σύμφωνα με τη μέρη διάταξη θα έχουμε τώρα δηλώσει Συμβουλίου και Επιτροπή, προετοιμασία τη συναντηση κορυφη κορυφής G7. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κατάινεν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο.